Η κυρία Πρόεδρο. Κυρίε και κύριοι συνάδελφοι, κυρία Επίτροπε, αρχίζει η συνεδρίαση. Καλή σα μέρα. Το πρώτο σημείο στην ημερήσια διάταξη είναι η έκθεση της κυρίας Μακάφη με θέμα